Καλησπέρα σας ε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται. Θέλω να σημειώσω ότι τα συνοπτικά πρακτικά της χθεσινής συνεδρίασης σας έχουν διανεμηθεί και αν δεν υπάρχουν παρατηρήσεις ε, θα θεωρήσω ότι τα πρακτικά εγκρίνονται. Η κυρία Χάρμς